Συνεδρίαση της Συνόδου Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η 22 Μαρτίου ήταν μια μαύρη μέρα για το Βέλγιο και μαύρη μέρα για την Ευρώπη. Ήταν η η τρομοκρατική αυτή επίθεση η οποία οδήγησε σε πολλούς θανάτους στις Βρυξέλλες. 32 αθώα άτομα έχασαν τη ζωή τους, 340 άτομα τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Αυτός είναι ο απολογισμός των αποτρόπαιων αυτών τρομοκρατικών ενεργειών που έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες, των απάνθρωπων αυτών τρομοκρατικών ενεργειών. Οι εγκληματίες του Ισλαμικού κράτους προσπαθούν με αυτές τις επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης να πλήξουν και τα ευρωπαϊκά όργανα και πολλούς άλλους θεσμούς της Ευρώπης με την επίθεση της Βρυξέλλες προσπάθησαν να χτυπήσουν τον πυρήνα της Ευρώπης. Την πόλη αυτή, την πολύγλωση, την κοσμοπολιτική, την ανεκτική πόλη που ενσωματώνει και εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή μας κοινότητα. Και η επίθεσή τους είχε σαν στόχο αθώα άτομα, αθώα άτομα, άτομα που τυχαία βρέθηκαν σε σημεία όπως το αεροδρόμιο ή το μετρό των Βρυξελών και πλήρωσαν με τη ζωή τους το γεγονός αυτό. Μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά, αυτό ήταν μια μορφή κοινικού υπολογισμού αυτών των τρομοκρατών. Θέλησαν με τον τρόπο αυτό όλοι οι πόλη των Βρυξελών όλο το Βέλγιο, όλη η Ευρώπη να καταληφθεί από ένα κλίμα τρόμου, ώστε ο φόβος να μπορέσει να μεταβληθεί σε μίσος. Γι' αυτό πρέπει να διατηρήσουμε τη διάβγειά μας. Δεν θα πρέπει να αφαιθούμε να περάσουμε σε μια γενική προκατάληψη και καχυποψία εναντίον των μουσουλμάνων και του Ισλάμ. Δεν πρέπει να εξισώσουμε το Ισλάμ με την διφλή βία. Θα πρέπει ως Ευρωπαίοι να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων, αλλά συγχρόνως να σταθούμε αλληλέγγυοι όλοι ως Ευρωπαίοι και να μην αφήσουμε να μας μολύνει ο φόβος που θέλουν να μεταφέρουν οι τρομοκράτες. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μίσος με μίσος, τη βία με βία. Δεν πρέπει να αφήσουμε να εξαπλωθεί μια υφέρπουσα μορφή καχυποψίας και φόβου προς άλλες κοινότητες. Θα πρέπει να κρατήσουμε τη συνεκτικότητά μας και με στόχο να εξασφαλίσουμε την ελευθερία όλων και τη δημοκρατία για όλους. Την αξία κάθε ανθρώπου. Και να τονίσουμε ότι αυτή είναι μια βασική αρχή που πρέπει όλοι να προασπίσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν σταθεί θύματα του τζιχαδισμού στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στο Ιράκ, στην ακτή του Ελφαντοστού, στην Τουρκία, στην Τινησία, Αίγυπτο, τη Συρία, τη Σομαλία, στην Ιγυρία, σε όλες αυτές τις χώρες, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν σκοτωθεί στους προηγούμενους μήνες εκατοντάδες αθώων ανθρώπων, που είναι τα θύματα αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Και ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης. Δεν θα πρέπει εμείς να ξεχάσουμε ότι αυτοί οι τρομοκράτες δρούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι μόνο Ευρωπαίοι, δεν είναι μόνο Μουσουλμάνοι. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μια απάντηση σε αυτή την τρομοκρατία. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατία σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την εσωτερική μας συνοχή και αλληλεγγύη. Όλοι μαζί, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ θέλω να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στα θύματα που έχουν τραυματιστεί και την πλήρη αλληλεγγύη μας θέλω να τονίσω με τις οικογένειες των αθώων θυμάτων των Βρυξελών. Έχουμε τα βαθιά συλληπιτήρια που θέλουμε να δώσουμε στις οικογένειες αυτών που έχασαν τη ζωή τους. Τα θύματα αυτά της τρομοκρατίας της Βρυξέλλες και σε άλλα μέρη του κόσμου δεν πρέπει να καλυφθούν από τη λύθη. Δεν, πρέπει, δεν έχουμε το δικαίωμα να τους ξεχάσουμε. Σας ζητώ λοιπόν να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή εις μνήμη των θυμάτων. Σας ευχαριστώ. Τα πρακτικά και τα εγκεκριμένα κείμενα από την προηγούμενη συνεδρία είναι στη διάθεσή σας. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις,